Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ελπίζω εφόσον ε, εσείς ασχολείστε και ε, του, ειδικά με τα θέματα του ανταγωνισμού στην ΙΜΚΟ και σας θέλω να σας ευχαριστήσω Νομίζω ότι από όλες τις ερωτήσεις ε, ένα πράγμα βγήκε σαν μήνυμα, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει ε, ε, τον ανταγωνισμό. Ένα ουδέτερο δίκαιο τρόπο εφαρμογής των κανόνων του ανταγωνισμού. Ταυτόχρονα δόθηκε και πώς η εφαρμογή του ανταγωνισμού θα διευκολύνει και θα βοηθήσει και άλλους τομείς ε, ε, οικονομικούς και πολιτικούς. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Σε κάποια από τα θέματα ίσως δεν στάθηκα πάρα πολύ συγκεκριμένη. Ελπίζω να επανέλθουμε, να τα ξαναπούμε. Ελπίζω να εκτιμήσατε ότι προσπάθησα να σας δείξω το ποιες είναι οι αξίες και οι αρχές τις οποίες πρεσβεύω. Και θα είναι η βάση της συνεργασίας για τα επόμενα πέντε χρόνια. Το μήνυμα από την συνάντηση αυτή, από την ακρόαση αυτή, είναι η δυνατότητα και η πίστη που έχουμε στον ανταγωνισμό που θα βοηθήσει τις περισσότερες επενδύσεις, την απασχόληση ε, και τις θέσεις απασχόλησης κυρίως. Ε, όλοι συνειδητοποιούμε επίσης το τι σημαίνει ε, η ψηφιακή οικονομία για τους πολίτες και εκεί θα πρέπει να υπάρξει ελεύθερος ανταγωνισμός και όχι κυρίαρχη θέση. Διότι είναι σημαντικό για τον καταναλωτή και για τον υπολογιστή λέει η υποψηφία επίτροπος. κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας μου εδώ έμαθα πάρα πολλά αρχικά. Μιλάμε για διάφορα αρχικά σε διάφορους τομείς. Και μετά έπεσα σε κάτι ρυθμίσεις για τον τρόπο με τον οποίο συναρμολογούνται τα παράθυρα και αναρωτήθηκα τι είναι αυτό, τι σημαίνει αυτό αποφάσεις για την συναρμολόγηση των παραθύρων. Ε, αφορούσε τα παράθυρα. Γιατί η παραγωγή ακριβώς ε, τέτοιου είδους κουφωμάτων ε, πράγματι ε, ήθελαν συγκεκριμένες προδιαγραφές και πράγματι υπήρξε μία απόφαση για τα κουφώματα των παραθύρων. Αυτό σημαίνει ότι πολλές εταιρείες προσπάθησαν ιδιαίτερα για να προωθήσουν αυτές τις απόψεις. Καταλαβαίνετε ότι μετά από μια τέτοια εμπειρία πώς ένιωσα. Αυτό το οποίο με βοήθησε πάντως είναι ότι η συνεργασία με σας πράγματι μπορεί να πάρει πολύ σημαντική, σημαντικό ρόλο. και μπορούμε να πετύχουμε πολλά, συνεργαζόμενοι και επίσημα και ανεπίσημα Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και όπως ε, είπα επανειλημμένα, ε, θα προσπαθήσω να πάρω μέρος σε αυτή τη μορφή συνεργασίας. Είμαι κόρη ιερέων στην εκκλησία της χώρας μου και μία από τις βασικές τους αρετές ήταν ότι καλωσόριζαν πάντα όσους έμπαιναν στην εκκλησία. Αντί να λένε άσχημα πράγματα για αυτούς που δεν έμπαιναν στην εκκλησία. Και γι' αυτό <laughs> καλωσορίζω όλους εσάς που ήρθατε εδώ σήμερα. Because I, I think it shows the dedication, which is actually and truly there. Αυτό δείχνει ακριβώς την αφοσίωσή σας στην υπόθεση αυτή. Και ελπίζω να είμαι ξεκάθαρη, θέλω να ευχαριστήσω τη διερμηνία, ελπίζω να διευκόλυναν αυτά τα οποία είπα την κατανόησή τους. Αγαπητά μέλη λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Ευχαριστώ Μάργαρετ Βέστακερ, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για την υπομονή. Τελειώνει εδώ η συνεδρίαση και σε 30 λεπτά έχουμε την αξιολόγησή μας και κλεισμένων των θυρών. Ευχαριστώ, πέρα συνεδριάσεως.